όλα τα εκκρεμή προβλήματα θα ε, βρουν μία λύση σε πνεύμα καλής θέλησης για να επιληθούν ταχύ. Ευχαριστώ εκ νέου. Αύριο στις 12. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο σημερινής διάταξη είναι η έκθεση της κυρίας ε, Ντελάνγκ, εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η εισηγήτρια, η κυρία Ντελάγκε, έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μέσω της έκθεσης αυτής ιδίας πρωτοβουλίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χτυπάει το καμπανάκι για την βιοπικιλότητα Νομίζω πως ε, τα είδη πεθαίνουν πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν. Μιλάμε για άνω από 30% των ε, αμφιβίων, 42% ε, των πτηνών και 52% των ψαριών του γλυκού νερού που απειλούνται με εξαφάνιση. Κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο όχι μόνο από βιολογική ή οικολογική σκοπιά, αλλά έχουμε και ηθική υποχρέωση να αφήσουμε πίσω τον κόσμο μας όπως τον βρήκαμε για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Και βεβαίως είναι και οικονομικά προς το συμφέρον μας να επενδύσουμε στην βιοπικιλότητα καθώς τα οικοσυστήματα μας ε, δίνουν καθαρό νερό, δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα κτλ. Οπότε η επιδείνωσή τους μας κοστίζει 50 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη δεν τα έχουν πάει καθόλου καλά εδώ πέρα. Επίσης δεν έχουμε επιτύχει και δεν είμαστε σε καλή πορεία για να επιτύχουμε τον ε, στόχο που είχαμε θέσει για το 2010. Ελπίζουμε όμως να τα καταφέρουμε για το 2020. Θα ήθελα όμως λοιπόν να κάνω κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις ε, συγκεκριμένες. Ε, θα πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με γωνίες και φέουδα. Η πολιτική της ε, φύσης θα πρέπει να αποτελέσει βεβαίως κομμάτι ολοκληρωμένων πολιτικών όπως η γεωργία, η αλληλεία, η περιφερειακή πολιτική και τα λοιπά. Βεβαίως έχουν γίνει τα πρώτα βήματα, το γνωρίζω, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτό τον δρόμο και βεβαίως μας δίνει την ευκαιρία αυτή η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής, π.χ. μέσω του να οργανωθεί μια κοινοτική υπηρεσία ε, για την αποζημίωση των αγροτών εκείνων οι οποίοι παράγουν με αηφόρο τρόπο. Επίσης να δημιουργήσουμε αμοιβαία υποφελείς καταστάσεις ε, εκεί όπου θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε και τις θέσεις εργασίας, πράσινες θέσεις εργασίας. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις περιοχές ε, Natura 2000 και για ένα ευνοϊκότερο καθεστώς τους. Βεβαίως η διαφορά που υπάρχει μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των ίδιων διατάξεων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επίσης ε, στηρίζουμε τις προτάσεις και τη φιλοδοξία της Κομισιόν όταν μιλάμε για την μείωση της υποχώρησης βιοπικιλότητας μέχρι το 2020. Είναι το ελάχιστο που θα πρέπει να έχουμε, αλλά και η αποκατάσταση της βιοπικιλότητας θα πρέπει να είναι κομμάτι της φιλοδοξίας μας και βεβαίως θα πρέπει να δούμε και σε διεθνές επίπεδο τι γίνεται. Οπότε θα πρέπει στη σύνοδο τη Εναγκόγια να πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να μιλήσει δυνατά και με μία φωνή. Θα πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να έχουμε κάνει τις μελέτες επιπτώσεων και τις οικολογικές και τις οικονομοτεχνικές. Όχι ως δικαιολογία αλλά για να είναι τα πράγματα ξεκαθαρία. Και τέλος ζητάω μια νέα πολιτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν μιλάμε ειδικά για τα ίδια εκείνα τα οποία είναι ξένα και εισβάλλουν σε ένα οικοσύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ενεργή διαχείριση χωρίς να υπάρξει αυτή η σωστή διαχείριση πλέον αυτών των οικοστημάτων δεν θα υπάρχει ε, καμία σωστή πολιτική. Εν φιλοδοξία και ρεαλισμό. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω του ε, σκιώδη ηγητέ για την ε, συνεργασία και για την ομόφωνη έγκριση τη έκθεση ε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Ποτότσνικο, ο οποίος βεβαίω δεν είναι εδώ γιατί είναι στη Νέα Υόρκη ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Ελπίζω όμως πως εφόσον μπόρεσε και ο κύριος Ντεχούφ να ακούσει αυτή την έκθεση στη μητρική του γλώσσα να του τα μεταφέρει. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της ε, Επιτροπής, ε, ο κύριος Δεούχτ για τρία uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, ο κύριος Ποτόσνικ τώρα που μιλάνε είναι στη Νέα Υόρκη για τις συζητήσεις στο ΝΟΙΕ για το Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι καταλαβαίνετε τους λόγους του οποίου δεν μπόρεσε να είναι παρόν εδώ. Για μένα λοιπόν, ε, σε, μένα μάλλον ανατέθηκε η απάντηση εξ ονόματος της Επιτροπής για την έκθεση της κυρίας Δελάνγκε, μια πολύ επίκαιρη έκθεση για την εφαρμογή της ευνοσιακής νομοθεσίας. Επίκαιρο είναι η σημαντική λέξη. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο σταυροδρόμι σε ό,τι αφορά την βιοπικιλότητα και την προστασία της φύσης. Η Επιτροπή συμφωνεί με τους βουλευτές ε, σε ό,τι αφορά την βαθιά ανησυχία μας για την ε, ταχεία απώλεια βιοπικιλότητας λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας ε, και την υποβάθμιση, την τρέπαστη υποβάθμιση πολλών, συστημάτων, πολλών οικοσυστημάτων που αποτελούν βασικό μέσο της επιβίωσής μας. Μετά την υιοθέτηση του στόχου του 2010 πετύχαμε κάποια πράγματα στην Ένωση για τα οποία μπορούμε να είμαστε περήφανοι το δίκτυο Natura 2000 ε, της Ένωσης επεκτάθηκε. Καλύπτει περίπου το 20% του εδάφους της Ένωσης και επεκτείνεται ακόμα και σε χερσαία και σε θαλάσσιες περιοχές. Η Ένωση προσπαθεί επίσης να επιτύχει τον ε, στόχο για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας μέχρι το 2010 παρά την τεράστια οικονομική κρίση στην Ευρώπη, υιοθετήσαμε το την περασμένη άνοιξη μια νέα οπτική για την βιοποικιλότητα. Οι νέοι στόχοι έχουν μεγάλη φιλοδοξία. Προσπαθούν, ε, ζητούν από την Ένωση να σταματήσει την υποβάθμιση ε, των τομέων της βιοποικιλότητας μέχρι το 2020. Ο πρόεδρος Μπαρόζο πρόσφατα ανέφερε στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης ότι η Επιτροπή θεωρεί πως αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα εξαιρετικής προτεραιότητας που πρέπει να αντιμετωπιστεί ταχύτατα. Ξέρουμε ότι ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι αντιμετώπισης ε, τη κατάσταση. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η ίδια φύση της πολιτικής ζωοπικιλότητας που είναι σύνθετη, καλύπτει τα πάντα. Η αποδοχή της ανάγκης ε, είναι αναγκαία, είναι, είναι, της αντιμετώπισης είναι βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του βασικού προβλήματος. Γιατί αλλιώ όλοι λένε φταίει ο άλλο και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Πρόκειται για μια εποχή μεταμόρφωση στην Ένωση πολλές πολιτικές με σημαντικό αντίκτυπο για τη βιοποικιλότητα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φάση αναθεώρησης. Τούτο συμβαίνει, για παράδειγμα, με την κοινή γεωργική πολιτική, την κοινή αλληλευτική πολιτική, την πολιτική συνοχή. Πρόκειται για. βρίσκονται σε σημαντικό. Βρισκόμαστε λοιπόν σε, μια, σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι ε, προσπαθώντας είτε να συνεχίσουμε την πολιτική προσπαθώντας να δώσουμε αποτελέσματα, είτε να αγνοήσουμε τους στόχους αυτούς λόγω των συγκυριών, αντιμετωπίζοντας πιθανές καταστροφικές επιπτώσεις. Το ψηφισμά μιλά πολύ για τις ανησυχητικές στάσεις απώλειας βιοποικιλότητας και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η τεράστια απώλεια και ο κίνδυνος οικοσυστημάτων και ειδών. Οι συνέπειες στην ε, ε, στα, στην αντιμετώπιση, στην επίτευξη των στόχων της χειριστίας. Η διαφύλαξη της ζωής στον πλανήτη είναι ένας βασικός στόχος που δεν πρέπει να, και δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει το μέγεθος της φιλοδοξίας αυτής. Επίσης η Επιτροπή ετοιμάζει μια ανακοίνωση για τη χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000 ε, προστατευμένων περιοχών, καλύτερη χρήση των εφιστάμενων πόρων και παροχή καλύτερης ε, ε, καλύτερων, περισσότερων ωφελιών στα ζητήματα βιοποικιλότητας. Συμφωνούμε με την έναση που η έκθεση δίνει για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας, χωρί την οποία δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε κανένα στόχο. Και περιμένουμε να κάνουμε περαιτέρω συζητήσεις με τα μέλη του Κοινοβουλίου για τα μέτρα πακέτο που θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε επιτυχώς τους νέους στόχους βιοπικιλότητας. Με την ίδια ευκαιρία θέλω να καλωσορίσω την εξαιρετική συνεισφορά ε, για την σχετική συζήτηση από την έκθεση της κυρίας Ντελάνγκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εκ μέρους της Επιτροπής η κυρία Λόβιν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ντελάνγκη για το έργο το οποίο επετέλεσε και με μεγάλη μας χαρά Εμεί τη Επιτροπή Αιλία μπορούμε να πούμε ότι συμφωνούμε και επιψηφίζουμε αυτήν την έκθεση που αποδεικνύει ότι 70 με 90% των ε, μεγαλύτερων ψαριών τώρα εξέλιπαν λόγω της υπεραλίευσης τα τελευταία 50 χρόνια. Άρα θα πρέπει να πάρουν να υπόθεση αυτή στα σοβαρά, διότι έτσι έχουν υπονομευθεί τα οικοσυστήματα στη θάλασσα που χρειάζονται για να απορροφάται το διοξείδιο του άνθρακα και για αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έτσι θα βοηθούσαμε και να σταματήσει η αλλαγή του κλίματος. Ε, είμαστε πρωτότυποι, ε, είμαστε πρωτοπόροι και στην Αγκόγια θα είμαστε επίσης για άλλη μια φορά στη διάσκεψη για το κλίμα. Οπότε εμείς ο πλευράς της Επιτροπής με μεγάλη μας χαρά διαπιστώνουμε ότι δόθηκε ιδέουσα σημασία σε έναν προγραμματισμό και σε μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη θάλασσα, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην διασυνδέονται οι επιμέρους πολιτικές μεταξύ τους. Άρα θα πρέπει να μπει ένα φρένο στην απώλεια της βιοποικιλότητας. Άρα θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά αυτή την υπόθεση και στα πλαίσια της πολιτικής της αλληλείας. Κύριο Σίμπερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ την κυρία Ντελάνγκη για την εξαιρετική έκθεση και τους κοιοδησίτες για την καλή συνεργασία. Τα στοιχεία είναι προφανή, περιέχονται στην έκθεση αυτή και είναι σαφές πως έχουμε ηθική υποχρέωση να διαφυλάξουμε τη βιοπικιλότητα αλλά και μια οικολογική και οικονομική υποχρέωση. Θα ήταν τρέλα λοιπόν το να μην είμαστε πιο επιτυχοί στο μέλλον. Ένα πρόβλημα βλέπω μόνο και αυτό είναι η αποδοχή των πολιτών. Και αν ε, μιλάμε και για το Natura 2000, διαπιστώνουμε πως σε κάποια κρατημέλη είναι πάρα πολύ επιτυχημένο, σε άλλα κράτη-μέλη όμως όχι τόσο και θεωρώ πως η Κομισιόν θα πρέπει να δώσει βάρος στο να μετράμε με το ίδιο μέτρο παντού. Δεν πειράζει κάποιους από ε, τους πολίτες το να υπερασπιζόμαστε την βιοποικιλότητα το αντιλαμβάνονται, αλλά δεν αντιλαμβάνονται το ότι κάποια κράτη σέρνουν τα πόδια τους ενώ κάποια άλλη είναι υπερβολικά αυστηρά. Εάν υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες ε, παντού νομίζω πως θα υπάρχει και πολιτική αποδοχή από το λαό κάτι το οποίο βεβαίως είναι εκ των όνων κάνευ για να επιτύχει αυτή η πολιτική και η Κομισιόν επιτέλους πρέπει να φέρει κατευθυντήρες γραμμές και εσείς βεβαίως ε, κύριε Πρόεδρε γνωρίζετε και εσείς ε, στην ε, χώρα σας πως υπάρχει ζήτημα με τη βιοποικιλότητα και μονίμως μας λέτε εμάς πως δεν μπορούμε να μετρήσουμε με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά για όλους. Ναι, κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ δεν θέλω τώρα να δείξω κάποια χώρα με το δάκτυλο. Το δάκτυλο απευθύνεται σε όλους μας γιατί η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2010 δεν λειτουργήσε οπότε θα πρέπει για τη νέα δεκαετία μέχρι το 2020 να βρούμε κάποιες νέες ιδέες. Βεβαίως σε λίγες εβδομάδες έχουμε τη διάσκεψη του ΟΗΕ για την βιοπικιλότητα στην Αγκόγια και νομίζω πως να μην είναι παρόμοια απογοήτευση όπως η διάσκεψη για το κλίμα στην Κοπενχάγη. Δεν επιτρέπεται να έχουμε πάλι αποτυχία σε μια τόσο σημαντική διάσκεψη για την προστασία της φύσης και έχει να παίξει σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση Νομίζω πως θα πρέπει να είμαστε υπέρ ενός φιλόδοξου προγράμματος ε, βιοπικιλότητας ε, και να δείξουμε αλληλεγγύη στη χρηματοδότηση αυτών των μέτρων και όπως είπαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μιλήσει με μία και με όχι με 27 διαφορετικές ε, φωνές. Αναφέρθηκε η έκθεση TIP 50 δισεκατομμύρια απώλειες ε, το χρόνο λόγω της απώλειας βιοποικιλότητας. Μιλάμε δηλαδή για ταυτόχρονα μια χρηματοδότηση η οποία είναι 0,2% για τη βιοποικιλότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματα δηλαδή τσιφούτικα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όσον αφορά την αλληλεγγύη μας με τον υπόλοιπο κόσμο χρειάζεται να μπορέσουμε και εμείς να προσφέρουμε κάτι ως αντάλλαγμα για τα είδη τα οποία παίρνουμε και εκμεταλλευόμαστε όταν μιλάμε π.χ. για τα ιατρικά φυτά. Χρειάζεται κάποιο είδου αποζημίωση σαν τις χώρες. Οπότε θεωρούμε πως είναι κάτι το εγκάρσιο η πολιτική της βιοπικιλότητας, γεωργία, αλληλεία, δασοκομεία, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε υπό το πρίσμα της ε, βιοπικιλότητας και βεβαίω υπάρχει και η οδηγία προστασίας ε, των εδαφών που αποκτάνε ο βάρος καθώς τα εδάφη βεβαίω αποτελούν ένα ανάχωμα, αν θέλετε, για το διοξείδιο του άνθρακα και θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ταχθεί υπέρ της βιοπικιλότητας και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ο κύριος ε, για Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεση Μία έκθεση βεβαίως η οποία ξεκινάει και μας λυπεί αυτά τα οποία αναφέρει για την αποτυχία της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής ε, από το 2000. Βεβαίως ε, όχι μόνο δεν επέτυχε αυτή η στρατηγική, ήταν γιγαντιαία αποτυχία. Δεν καταφέραμε να μειώσουμε το ρυθμό μείωσης ε, καν και φαίνεται πως η πείνα μας αυτή δεν ε, μπορεί να κορεστεί με τίποτα και καταβροχτίζουμε τον πλανήτη. Βεβαίως θα πρέπει να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Βλέπουμε λοιπόν πως ε, έχουμε ένα κατάλογο απειλουμένων ειδών που αυξάνεται και έχουμε πολύ καλές δηλώσεις, ωραίες δηλώσεις από την άλλη μεριά του Συμβουλίου προς τον ε, ΟΗΕ, αλλά αν δούμε τι γίνεται όταν πρέπει δηλαδή πραγματικά να πονέσουμε και να γίνουν επιλογές, τότε υπερισχύουν πάντα τα συμφέροντα των, ψαρό, των ψαράδων, των αγροτών, της δασοκομείας. Κύριε Πρόεδρε, μας λένε οι μελέτες ε, πως ε, οι λανθασμένες αυτές ε, επιλογές θα μας κοστίσουν 7 10% του ΑΕΠ, 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για πάρα πολλά μηδενικά το έτος. Οπότε θα πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα όταν χαράξουμε τη νέα πολιτική για τη γεωργία, για την αλληλεία, τις νέες εμπορικές συμφωνίες που κλείνουμε. Θα πρέπει λοιπόν και οι υπουργοί οι ίδιοι που κάνουν όλες αυτές τις ωραίες ε, δηλώσεις να κάνουν και τις σωστές επιλογές. Αλλιώς η στρατηγική αυτή θα είναι ένα κομμάτι χαρτί όπως και η προηγούμενη. Και βεβαίως αυτή η χάρτινη, χάρτινη στίγρηση αντίστοιχη με τις πραγματικές από ό,τι φαίνεται δεν θα εξαφανιστούν ποτέ. Η κυρία Μπελιέ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως αναφέρθηκε, φέτος είναι το Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας. Φέτος λοιπόν είμαστε, σε έχουν καλέσει να αντιμετωπίσουμε μια τριπλή κρίση που, συνδέεται μεταξύ τους και απαιτεί μια ε, ενοποιημένη προσέγγιση για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Την οικολογική κρίση που έχει συνέπεια και στην ε, κοινωνική οικονομία και την κοινωνία. Ε, επισητιστική ε, ασφάλεια, βιοκλιματική και απώλεια βιοποικιλότητας. Να υπενθυμίσουμε ότι δεν υπάρχει τίμημα για τη βιοποικιλότητα. Οδηγεί ωστόσο σε αύξηση της φτώχειας, δημιουργεί σοβαρές ανισοδοποίες οικονομικού χαρακτήρα, ευημερίας, αλλά και ανισοδοποίες πολιτισμικού χαρακτήρα, όπως ένα αναφέρθηκε, το 40% της παγκόσμιας οικονομίας εξαρτάται ε, από τις υπηρεσίες που παρέχει η φύση. Το 60% αυτών βρίσκεται σε παρακμή. Η Ευρώπη έχασε το 40% της βιοπικιλότητάς της τα τελευταία χρόνια. 50 δισεκατομμύρια το χρόνο έχει κόστος αυτή η έλλειψη. 14-3 το 2050 θα φτάσουν οι ζημιές αν δεν προχωρήσουμε, διότι τα φαινόμενα επιταχύνονται και ε, οι, οι λόγοι είναι γνωστοί. Τους αναφέρει και η έκθεση. Τα μέτρα επίσης αναφέρονται στην έκθεση. Ελπίζουμε να υπερψηφιστεί ευρέω η έκθεση αυτή και ευχαριστούμε την κυρία Ντελάνκη και τη δουλειά τη. Ωστόσο, πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις, από τις συζητήσεις στους στόχους και να υπογραμμίσουμε την μικρή αντίδραση του Συμβουλίου και της ε, επιτροπής. Η οδηγία για το νερό και για το έδαφος έχει μείνει στις συζητήσεις. Ε, είναι, είναι λυπηρό το ότι δεν υπήρξε μεγαλύτερη ένταξη της βιοποικιλότητας στη γενικότερη στρατηγική της Ένωσης την, ένταξη του οικολογικού εμπορίου στην οικονομία μας. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια και να καταλάβουμε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε την διαφύλαξη και την ανάδειξη του κεφαλαίου σε φύση. Αυτό είναι μια επένδυση που οδηγεί σε κέρδη για το μέλλον. Κύριε Πρόεδρε, διαπιστούμε πως ε, το έτος 2010, το έτος βιοπικιλότητας, ε, δεν έχουμε επιτύχει τους ε, στόχους. Έχουμε λοιπόν λόγους για σοβαρή ανησυχία. Μιλάμε για τον πυρήνα της δημιουργίας ε, του παντοδύναμου. Μιλάμε για την ε, βάση των ε, τροφίμων που χρειαζόμαστε και τη γεωργίας και βέβαια συνεισφέρει σε ένα σταθερό κλίμα. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσει η απώλεια της βιοποικιλότητας και να αναλάβουμε συγκεκριμένη δράση. Πρέπει λοιπόν Κομισιόν, Κοινοβούλιο και κράτη-μέλη να μιλήσουν με μία φωνή να θέσουν φιλόδοξους στόχους για την επόμενη δεκαετία για να σταματήσει η απώλεια βιοπικιλότητας, να υπάρξει ένα παγκόσμιο όραμα για την προστασία των οικοσυστημάτων και την αποκατάστασή τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερέιρα για ένα λεπτό. Obrigado, Sr. Presidente. A definição de uma rede ecológica coerente à escala europeia que reúna hábitats relevantes e representativos. Κύριε Πρόεδρε, τον έχουμε ένα τέτοιο δίκτυο και έτσι να έχουμε αυτούς τους δεδομένους τόπους σε ένα δίκτυο είναι ένα, μια, ε, ένας μόνο παράγοντας ε, να διασώσουμε την βιοποικιλότητα. Όμως θα πρέπει να έχουμε κάποιους παράγοντες ούτως ώστε να μπορούμε και τις απειλές να ελέγξουμε αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε πέρα από αυτό να ανακτήσουμε ό,τι έχει επιδεινωθεί, ό,τι έχει χαθεί. Οπότε δυστυχώς ε, ένα τέτοιο δίκτυο που είχε γίνει με τον Αντρόεδρο 2000 δεν συνοδεύτηκε από επιστημονικά μέτρα ε, και γι' αυτό το λόγο δεν ήταν αποτελεσματικό το Natura 2000. Επίσης, οι περικοπές που έγιναν δεν ήταν σωστές. Ε, ε, ό,τι προβλέπει δηλαδή ο προϋπολογισμός του 2010, ενώ προβλέπει αυξήσεις στρατιωτικών δαπανών. Επομένως, θα πρέπει τώρα να δούμε πώς θα μπορέσουμε αυτή την υπόθεση να την εντάξουμε και σε άλλες τομιακές πολιτικές και γι' αυτό και θα πρέπει να προχωρήσουμε ε, σε μια προσαρμογή των αντιστοίχων ε, πολιτικών της ΚΑΠ, της συμπορικής πολιτικής και άλλων. Ε, ο κ. Ντεφίχτη, ο οποίο είναι ο κυρίω αρμόδιο με το χαρτοφυλάκια ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να κάνει τη χρήση για να σωθεί δύο Ρόσπαχ, Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς έχουμε ενώπιόν μας σήμερα μια τέτοια χτιστική πιλότα που λέει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι η κοινή αλληλευτική πολιτική θα πρέπει να βοηθάει στη τους του θα πρέπει να γίνουν αναγκαίε αλλαγέ. Και το ίδιο ισχύει και για την ΚΑΠ. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την παλαιότερη πολιτική, τα λοιπάσματα και τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούσαμε. Να γίνουμε ανταγωνιστικοί στη παγκόσμια σκηνή, αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε και το περιβάλλον. Βιομηχανία, αλληλεία και γεωργία θα πρέπει να συμμορφωθούν. Όλοι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει όλα αυτά τα οποία λέμε να βοηθήσουν να γίνουν πράξη. Η κυρία Γκουτιέρες για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η χρονιά αυτή αφιερωμένη στη βιοπικιλότητα ε, πέρασε με λίγες λύσεις και πολλή κουβέντα για την τραγωδία περνάμε ενώ η κοινωνία χρειάζεται λύσεις νέες μορφές προσέγγισης στο πρόβλημα πρώτα-πρώτα ε, αυτό το οποίο έγινε όσον αφορά την κατανομή σε γεωγραφικές ζώνες θα πρέπει να συνοδευτεί από συγκεκριμένη πολιτική γιατί ε, η κάθε περιφέρεια έχει τα δικά της προβλήματα στην Ευρώπη άρα να κάτσουμε και να επεξεργαστούμε μια μικροπολιτική ε, συγκεκριμένη σε, στην τοπική σφαίρα αυτό χρειάζεται η βιοπικιλότητα το έδαφος, η απερίμωση των ε, γεωργικών γεών, ε, όλα αυτά τα έχουμε αφήσει. Θα πρέπει όμως ε, ακόμα και το, και το τι τρώνε τα ζώα πρέπει να το φροντίσουμε ανάλογα με την κάθε περιφερεια γιατί το θέμα δεν είναι τι γίνεται με τα πουλιά και τα ζώα σε κάθε περιοχή αλλά το θέμα είναι και το τι γίνεται και με τα έντομα γιατί λείπουν τα έντομα, χάνονται και να γιατί έχουμε απόλυτη ποικιλότητα, γιατί έτσι δεν έχουν να φάνε τα πουλιά και πάνε και τα πουλιά. Άρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την οργανική σύσταση του, του εδάφου και αυτό το οποίο κάνουμε τώρα είναι ένα πανευρωπαϊκό έγκλημα επίση. Ε, οι γεωκτήμονε είναι σημαντικό ε, παράγον. Ε, κάναμε μια επιτροπή, εγώ εκεί είναι όλοι εμπλεκόμενοι, όμω ε, τι γίνεται με, με τον ε, Γιώργο. Ο Γιώργος φυτεύει αυτά τα οποία εμείς ε, τρώμε και ο, και ο, και ο γεωκτήμων. Επομένω, δεν θα πρέπει δικτατορικά να επιβάλλουμε ιδεολογικέ πλατφόρμε. Θα πρέπει αυτό να λάβει τέλο και μόνο έτσι θα μπορούμε να σώσουμε τη διοπικιλότητα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είπε η κυρία Ντελάνγκη ότι χτυπάει το καμπανάκι. Όντω έτσι είναι. Αλλά χτυπάει ταυτόχρονα και η απογοήτευση όπως ακούγεται διότι δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι της ηλιετίας. Αυτά που διακυβεύονται είναι πολλά. Ο φυσικός μας περίγυρος είναι τόσο τροτός που καταλαβαίνουμε ότι ό,τι δεν πληρώσουμε τώρα, θα το πληρώσουμε από την, ε, το πορτοφόλι των γενεών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πολλά για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, παίζοντας ε, και χρησιμοποιώντας μια σειρά μέτρων. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις η αποτυχία δεν οφείλεται σε, σε ε, έλλειψη ικανότητας, αλλά σε αδυναμία, σε έλλειψη βούλησης. Η βιοπικιλότητα δεν είναι κάτι ε, ένα μουσιακό, ε, μια μουσιακή έκθεση που πρέπει να την κλείσουμε και την διαφυλάξουμε. Η βιοπικιλότητα υπάρχει παντού. Δεν γνωρίζει, ε, δεν γνωρίζει σύνορα. Χρειάζεται να υπάρξει μια παγκόσμια βούληση, όχι μόνο κοινοτική, ιδίω σε ό,τι αφορά το έδαφος. Η επικουρικότητα σαν, μέσο, σαν μόνο εργαλείο αντιμετώπισης της υποβάθμισης του εδάφους, ιδίως στα δάση, μπορεί να αποτελέσει ένα νέο μέσο ε, ένα δεύτερο θέμα. Μια κοινή πολιτική στην προστασία του εδάφους θα έχει θετικές συνέπειες στην Ευρώπη που είναι τόσο διαφοροποιημένο αλλά που, θα δείχνει, που δείχνει ταυτόχρονα την έλλειψη βούλης των κρατών μελών και την έλλειψη πραγματικής ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στον τομέα του εδάφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ντελάνκια για την έκθεσή της για την ευρωπαϊκή βιοπικιλότητα. Η Ευρώπη δεν καταφέρνει να σταματήσει την απώλεια βιοπικιλότητας και αυτό είναι κάτι το σημαντικό και δικαίως η κυρία Ντελάνκη ζητάει να δώσουμε προσοχή και εμείς στηρίζουμε την ε, Κομισιόν και την προσπάθειά της να σταματήσει τουλάχιστον το 2020 η απώλεια της βιοπικιλότητας. Αυτό σημαίνει λοιπόν πως θα πρέπει να αλλάξει η γεωργική πολιτική, να αλλάξει η πολιτική αλίας, να αλλάξει η πολιτική υποδομών, να αλλάξει η περιφερειακή ανάπτυξη, όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε την επόμενη περίοδο στις δημοσιονομικές προοπτικές και υποθέτω πως η κυρία Ντελάνγκε και Φαντάλε που είπαν τόσο καλά λόγια για τη βιοπικιλότητα θα τα μεταφράσουν αυτά τα πράγματα και σε δημοσιονομικές προοπτικές εάν πραγματικά θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή την πολιτική. Αλλιώς μιλάμε για ένα αποκάμισο αδιανό. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, υπάρχει γενικότερη αναγνώριση του ρόλου των γεωργών στην διαφύλαξη της ε, και στις καλές πρακτικές. Συζητούμε τώρα τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής και ένα από τα βασικά εργαλεία, ένα από τα βασικά επιχειρήματα ε, είναι η υπεύθυνη ε, γεωργία και ο τρόπος αποζημίωσης των υπεύθυνων γεωργών καθότι παρέχουν ένα δημόσιο αγαθό. Πιστεύω ότι δεν, ε, ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση αυτή. Θα πρέπει οι γεωργοί να προωθήσουν ε, αγρο, αγροτικά, αγρο, αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και να λειτουργήσει περισσότερο σαν καρότο η προσέγγιση αυτή και όχι ως ε, μπαστούνι. Μίλησε η κυρία Ντελάγκη για, την ιδιότητα, για, για μια σειρά ενδιαφερουσών ιδεών που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν συμφωνώ με όσους λένε ότι πρέπει να αλλάξει οδηγία. Χρειάζεται εμένα, αλλά υπάρχουν επαρκή εργαλεία πριν γίνει κάτι τέτοιο και νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ε, που αντιμετωπίσουμε μέχρι τώρα. Ε, δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει ωστόσο με την υφιστάμενη μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ από πλευρά μου συγχαρώ την εισηγήτρια, την κυρία Ντελάγκε, για το έργο της. Για να μπορέσουμε να διασώσουμε το οικοσύστημα, το κλίμα, την ατμόσφαιρα, το έδαφος, τα τρόφιμα, θα πρέπει να προστατεύουμε τη βικιλότα και άρα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, τόσο ώστε αυτό το κεφάλαιο να περισσωθεί, ούτω ώστε να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και άρα θα πρέπει να δούμε πώς με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα προστατεύσουμε το περιβάλλον και έτσι θα έχουμε οικολογικές λύσεις. Τα καλά νέα είναι το live τώρα θα έχει καλύτερη πρικοδότηση έστω και κατά ο λίγο. Χρειαζόμαστε επομένω καλύτερε, μεγαλύτερε επενδύσει και αυτή είναι η προστιθέμενη αξία για την πόση βιοπικιλότητα. Και άρα θα πρέπει να αποθαρρύνουμε τι επενδύσει που είναι κατά τη βιοπικιλότητα και από δημόσιο και από ιδιωτικό τομέα. Και γι' αυτό καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη όλες τις μεταβλητές για να έχουμε μια βιώσιμη πολιτική που να είναι υπέρ του περιβάλλοντος. Ehm, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούγοντας τους συναδέλφους βλέπω πως υπάρχει συνένεση για το κατεπήγον του πράγματος, ε, αλλά πρέπει να πάμε στην ουσία του πράγματος. Το πρόγραμμα περιβάλλοντος του ΟΗΕ υπολόγισε πως η επένδυση στη βιοπικιλότητα μπορεί να αποδώσει. Κάθε ευρώ μπορεί να αποδώσει ε, από 3 μέχρι 75 φορές ε, την αξία του. Οπότε υπάρχει και οικονομική αξία, αλλά πρέπει να το δούμε αυτό σε όλους τους τομείς μας, δηλαδή αλληλεία, γεωργία και τα διαρθρωτικά ταμεία. Όσον αφορά τη γεωργία, βλέπουμε πως υπάρχουν κάποια, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο στην προώθηση της βιοπικιλότητας δεν είναι μόνο το LIFE, ε, πρέπει να ενταχθεί σε όλους τους δυνατούς ε, τομείς ε, στους οποίους δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τον βλέπω. Η κυρία Φράγα Εστέβες για 1,5 λεπτό είναι εδώ. Δεν την βλέπω. Η κυρία Καρβάλιο για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, είναι σημαντική αυτή η έκθεση γιατί θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο να βρούμε τη βιοπικιλότητα. Δυστυχώ όμω, ο στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που το Γκέτεμπορκ κύρωσε το 2001 δεν υλοποιήθηκε. Και οι συνέπειε είναι ότι έχει υποθηκευτεί το μέλλον μα, η ευημερία μα. Και άρα θα πρέπει να δούμε και ότι υφιστάμεθα και συνέπειες οικονομικές. Το Natura 2000 είχε κάποιους συγκεκριμένου στόχους. Οπότε θα πρέπει να ζητήσουμε τα κράτη-μέλη να δώσουν προτεραιότητα όσον αφορά την υλοποίηση του Natura 2000. Επίσης είναι σημαντικό να εντάξουμε τη βιοποικιλότητα και σε άλλες πολιτικές, γεωργία, τουρισμός, ε, ανάπτυξη υπαίθρου, αλία και αντίστοιχα θα πρέπει να φροντίσει και ο προηγούμενος να καλύψει κάποια επιστημονική έρευνα για την βιοπικιλότητα και να βοηθήσει και το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Και για όλους αυτούς τους λόγους είναι θετικό το ότι έχουμε τώρα κεντρική προτεραιότητα τη για το 2020. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, περνάμε τώρα στη διαδικασία του ΚΑΣΤΙΑΗ. Ο κύριος Κέλλη για ένα λεπτό. Ε, thank you, Mr. President. Ε, Ευχαριστώ. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει όλα τα, όλα τα πλάσματα του Θεού είναι, μεγάλα και μικρά. Κάποια από τα μικρά πλάσματα αρχίζουν και χάνονται, κυρίως λόγω της δουλειάς των μεγάλων πλασμάτων, του ανθρώπου κυρίως, του Homo sapiens. Είναι καιρός λοιπόν να, να μπει λίγη λογική στη συζήτηση αυτή. Ε, μίλησα με την κύριε Ντελάγκη και άλλους ομιλητές. Ο χρόνος τρέχει εις βάρος μας. Τα οικονομικά επιχειρήματα είναι ξεκάθαρα. Μια ζήλια 40-50 δις απολειών ε, που αν δεν αντιμετωπιστεί τώρα θα φτάσει στα 14-3 σε λίγα χρόνια. Ο κύριος Νίκο, κύριε Νίκολσον, ε, καλά είναι τα καρότα προς τους γεωργούς και τους ε, ψαράδες, αλλά καλή είναι και η εκπαίδευση. Εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση. Ο κύριος Σόνικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε πως το 2010 θα πρέπει να είναι το έτος βιοποικιλότητας. Οπότε πρέπει να γίνει μια παγκόσμια εκστρατεία ενημέρωσης για την προστασία της βιοποικιλότητας. Όμως, ε, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, μόνο 38% των Ευρωπαίων ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Οπότε πρέπει να δούμε τι έχουμε επιτύχει όσον αφορά λοιπόν τη βιοπικιλότητα. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να σταματήσουμε την απώλεια της βιοπικιλότητας. Έχουμε τις λεγόμενες ημέρες κληρονομιάς ε, που κυρίως ε, βεβαίως αφορούν την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Ίσως η Κομισιόν θα έπρεπε να οργανώσει κάποιες μέρες κληρονομιάς βιοπικιλότητας. Επίσης, η διάσκεψη της Ναγκόγια πλησιάζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ εγώ πως θα πρέπει να έχει σαφή θέση για την προστασία της βιοπικιλότητας πέρα από το 2030. Είτε μιλάμε για χρηματοδότηση, είτε για κοινέ δράσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να δούμε προσεκτικά και με αηφόρο τρόπο το μεγάλο δώρο που μας έχει κάνει η φύση και να το εκμεταλλευτούμε σωστά το να εκμεταλλευτούμε ε, τη φύση και τους αγρούς βεβαίως δεν είναι καμία αντίφαση αυτό φαίνεται και στην ε, πατρίδα μου όπως ε, παραδείγματο χάρη σε ορισμένα αμπέλια στα οποία γίνεται αγρανάπαυση έχει επιστρέψει ένα σπάνιο είδος πεταλούδας και βλέπετε πως υπάρχει και η δυνατότητα από ορισμένα φυτά να ανακαλυφθούν νέες θεραπείες και νέα φάρμακα και θα πρέπει να υπάρξει και μία ανάλογη βεβαίως αποζημίωση. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω μιας νέας κοινή γεωργική ε, πολιτική. Νομίζω κάποια επίση από τα προγράμματα μας πρέπει να επανεξεταστούν και διαπιστώνουμε πως οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε λοιπόν περαιτέρω υποχρεώσεις αλλά και ενιαίους ελέγχους όσον αφορά δε, την προστασία των εδαφών ε, μπορούν να το κάνουν και τώρα τα κράτη-μέλη δεν χρειάζεται να περιμένουμε και άλλη ευρωπαϊκή οδηγία ευχαριστώ Ευχαριστώ την κυρία Ντελάνγκε διότι μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια πολλοί Ούγγροι γεωργοί υπέβαλαν ε, παραπονέθηκαν μάλλον λέγοντας ότι θα μείωναν, ε, ότι θα μείωναν τα οι που θα λάβαιναν αν δεν έκοβαν δέντρα και θάμνους. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε από μια μεριά και πληρώνουμε για να δημιουργήσει κάποιος έναν φυσικό βιότοπο για πουλιά, από την άλλη υποστηρίζουμε και χρηματοδοτούμε το κόψιμο δέντρων και θάμνων. Δεν γνωρίζει η αριστερά τι πει η δεξιά που λέει και η γεγραφή. Κλασικό παράδειγμα των προβλημάτων στην μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε τώρα που συζητούμε τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και να σκεφτούμε πού πρέπει να δοθεί η προτεραιότητα, στη βιοπικιλότητα. Πρόεδρε, επίτροπε, πολύ σημαντική έκθεση. Συγχαρητήρια για την εισηγήτρια και θέλω να μιλήσω για ένα βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ε, ε, οικοσυστημάτων. Το Natura 2000 που καλύπτει 20% του χερσαίου εδάφους της Ένωσης, 17% του ε, της στη Ρουμανία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιτροπής, το ετήσιο κόστος διαχείρισης των δικτύων Natura 2000 ανέρχεται σε 6,5 δις ευρώ. 242 εκατομμύρια για τη Ρουμανία. Πρέπει να πετύχουμε τους στόχους αυτούς, άρα πρέπει να προστατεύσουμε την βιοπικιλότητα. Διαπιστώνω ότι η Επιτροπή πρέπει να δώσει συμπληρωματικά κονδύλια για την προστασία της βιοπικιλότητας. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο κάνοντας και μια ενδιάμεση αξιολόγηση του δημοσιονομικού πλαίσιου 2007-2013 γιατί δεν έχουν πετύχει τους στόχους του 2010. Ευχαριστώ. Επίτροπε συνάδελφοι, η διαφύλαξη της βιοπικιλότητας είναι σημαντικό ζήτημα, επίκαιρο ζήτημα. Υποτιμάται από πολλούς ωστόσο. Μέγα τμήμα των πολιτών στα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης δεν καταλαβαίνουν το σοβαρό κίνδυνο που σημαίνει η μείωση της βιοποικιλότητας ούτε τις συνέπειες που κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει το κλίμα, το περιβάλλον και τις οικονομίες των χωρών. Είμαι βέβαιο ότι η δική μας αρμοδιότητα είναι να υλοποιήσουμε απόλυτα την υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία, να ενσωματώσουμε χρηματοδότηση στις πολιτικές για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και να απλοποιήσουμε κανόνες για την πρόσβαση και τη χρηματοδότηση σε σε τοπικά έργα όπως το πρόγραμμα LIFE που ανέφερε ο συνάδελφος Αντωνέσκο. Τη διαφύλαξη των ε, θαλάσσιων και χερσαίων οικοτόπων πρέπει να είναι προτεραιότητα όχι μόνο τον, της Ευρώπης αλλά και των κρατών μελών που θα πρέπει να, ενημερ, να ενημερώνουν όσους παθαίνουν να παρεμβαίνουν και τα κάθε επίπεδο, τοπικό και άλλο, για τα κριτήρια διαφύλαξης της βιοποικιλότητας. Κλείνω υπενθυμίζοντας ότι το Κοινοβούλιο έχει την ευθύνη να δώσει σαφές μήνυμα προς την υπόλοιπη Ευρώπη για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας, ιδίως δε τον, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των επερχόμενων γενεών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ακούσω τον κόνδυνα του κινδύνου σε σχέση με τα όσα μας λέει αυτή η έκθεση. Κατόπιν και σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες είπαμε ότι η εθνισμότητα στη Μαύρη Θάλασσα όσον αφορά τα ψάρια όλο ένα και αυξάνεται και στο Δνύστερο αλλά και στον Δούναβη στα ποτάμια μας υπάρχει τόσος φόσφορος που μολύνει και άζωτο και άλλες οργανικές ουσίες που όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια τεράστια απειλή για τα ψάρια. Άρα το πρόβλημα αυτό να θεωρηθεί η ψήστη προτεραιότητα στην μέση διάταξη της Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό και θέτω πολύ θετική σημερινή έκθεση και συγχαρητήρια προς την κυρία. για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την κυρία Ντελάνγκη για την εξαιρετική της έκθεση και βεβαίως η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική αλλά νομίζω πως εδώ πέρα μας διαφεύγει κάτι σημαντικό οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί που είναι μια τεράστια απειλή για την ε, βιοπικιλότητα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη δεν έχουμε βεβαίως τόσο πολλές καλλιέργειες γενετικά τροποποιημένων οργανισμών αλλά συνεχώς ε, υφιστάμεθα πίεση για να επιτρέψουμε την καλλιέργειά τους και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό για την γεωργία. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο με μεγάλη παραγωγή και μονοκαλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, είμαι σίγουρος πως το τίμα το οποίο θα πληρώσουμε θα είναι η απώλεια βιοπικιλότητας. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσπαθήσει να υπερασπιστεί εαυτόν και πολιτικά, γιατί ξε, βεβαίως ξέρω και τις τοποθετήσεις διαφόρων πολιτικών ομάδων, οπότε είναι δύσκολο να έχουμε πανευρωπαϊκή απαγόρευση, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να μην υπάρχουν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις σε σοδιές ε, τέτοιες. Δεν είναι ανάγκη να το επιδοτούμε και με ευρωπαϊκά κονδύλια. Σας Αξιότιμοι συνάδελφοι, η βιοπικιλότητα μας αφορά όλους. Πρέπει να έχουμε ενιαίες οδηγίες γιατί το πρόβλημα της καταστροφής των οικοσυστημάτων και της απώλειας βιοπικιλότητας δεν σταματάει στα σύνορα. Οπότε συμφωνώ και εγώ εδώ πέρα και συντάσσομαι με την έκκληση οι Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να έχουν κοινέ δομέ αποφάσεων και να βελτιώσουν και τις ε, διαχειριστικές δομές.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 Είναι μία εξέλιξη τριών χιλιάδων ετών η οποία επέτρεψε να προσαρμοστεί η ζωή και οι μηχανισμοί της προς το μέλλον και αυτό είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της εξέλιξης αλλά επίσης και ένας τρόπος με τον οποίο όλες οι γεννητικές και μορφολογικές αλλαγές μπορεί να καταλήξουν σε νέα είδη. Η βιοπικιλότητα είναι μία ε, πολιτική η οποία εξασφαλίζει την διαιώνιση των ειδών και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την διατηρήσουμε, για να μειώσουμε τις κλιματολογικές αλλαγές, να μελετήσουμε, να έχουμε τις ουσιώδες γνώσεις και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ε, την, ε, ε, τις ιατρικές εφαρμογές της πανίδας και της χλωρίδας. Ο κύριος Ντεγκούχτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να απαντήσω σε μερικά ουσιαστικά θέματα και μετά να κάνω καταληκτικές παρατηρήσεις. Όσον αφορά τους κοινού κανόνες για την βιοπικιλότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη και τους ενδιαφερόμενους για να επεξεργαστεί κατευθυντήριες γραμμές στους διάφορους τομείς που μας απασχολούν και στα πλαίσια του προγράμματος προγράμματος Natura 2000. Η νέα στρατηγική βιοπικιλότητος θα εστιαστεί στην ενίσχυση της ε, ολοκλήρωσης των πολιτικών που επηρεάζουν την πολιτική, ε, την γεωργική, της ε, αλληλείας και θα προσπαθήσει να επιτύχει τους στόχους που θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα τη στρατηγική του 2020 και που αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά την προστασία του εδάφους, ε, προτείνουμε να υπάρξει ε, ένα ε, κείμενο το οποίο θα απαντήσει εις τις ανησυχίες σας για την επιδείνωση της κατάστασης των εδαφών και θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση σε συνεννόηση με το Συμβούλιο. Και τέλος θα ήθελα να σας πω ότι είναι καλό να αντιλαμβάνεται κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συμμερίζονται τις ίδιες ανησυχίες σχετικά με την διατήρηση του οικοσυστήματος και θα πρέπει να κοιτάξουμε να επιτύχουμε τους στόχους της βιοπικιλότητος που κατευθυνθήκαν το 2010 και το 2000 2020 να μην ε, χρειαστεί να αποδεχθούμε ότι αποτύχαμε και δεν ε, διατηρήσαμε τη βιοπικιλότητα στην Ευρώπη. Και ολοκληρώνω με το σλόγγαν μας για το τρέχον έτος, το έτος της βιοπικιλότητας ότι είμαστε όλοι μαζί και μόνο μαζί θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον πλανήτη για να επιτύχουμε την ποικιλομορφία ζωής και ε, θα δώσω το, θα έδινα το λόγο στον κύριο Ποτόσνικ αλλά όπως γνωρίζετε είναι στη Νέα Υόρκη ε, για ένα πολύ σημαντικό συνέδριο σχετικά με αυτό το θέμα και γι' αυτό τον καθιστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις διάφορες προοπτικές που μας προσέφεραν. Όλες οι παρεμβάσεις επεσήμεναν τη σημασία της ε, διεθνούς ε, θέσης για το mainstreaming και ο Επίτροπος θα πρέπει να το συμπεριλάβει αυτό στη στρατηγική του. Θα πρέπει να προσδώσει την απαραίτητη ε, σαφήνεια για να υπογραμμίσει τα θέματα ε, που είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ των. για τις προθεσμίες ακούσαμε όσα έπρεπε να ακούσαμε και θα πρέπει πράγματι να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Η πολιτική της αλληλείας ε, και οι διάφορες δομές αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων και θα ήθελα να απαντήσω στους συναδέλφους και να τους πω ότι το mail stream αναφέρεται και στη χρηματοδότηση. Δεν έχει σημασία για μένα από πού προέρχεται η χρηματοδότηση. Αυτό που έχει σημασία είναι να είναι αποτελεσματική η χρηματοδότηση. Και ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πιάσουμε με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Να έχουμε ω ως στόχο μία ενιαία χρηματοδότηση. Ήταν μια ανοιχτή ερμηνεία αυτή τη παροιμία, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να προσπαθήσουμε να πιάσουμε τρία ή τέσσερα τριγώνια με τον ίδιο σπάρο. Επομένω, λοιπόν, ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το, σύστημα, το θέμα αυτό σε διεθνέ επίπεδο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο συνάδελφο Ροντρίγκε αναφέρθηκε σε μια ομοιόμορφη διαχείριση του εδάφους ε, στην Ευρώπη εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πόσο διαφορετικό είναι το έδαφος στη διάφορα σημεία του κόσμου και επομένω είναι απαράδεκτο το όλο θέμα του εδάφους ε, για παράδειγμα στην Ολλανδία που εμείς έχουμε έδαφος τρία μέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας είναι τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση που θα έχουμε σε μια άλλη χώρα που είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση. Ε, δεν μπορούμε βέβαια να μιλάμε μόνο για αρμοδιότητε για χρηματοδότηση και να ξεχνάμε τις παρεμβάσεις. Θα πρέπει να υπάρχει δημόσια διαχείριση και αρχές. Δεν αναφερθήκαμε επίσης ε, και στις ε, δεσμεύσεις των επιχειρήσεων. Αν θέλουμε να γίνουν πραγματικά βήματα προς το μέλλον, δεν θα πρέπει να σκεφτούμε μόνο τις δημόσιες αρχές, αλλά να σκεφτούμε και όλες τις υπόλοιπε πτυχές. Ευχαριστούμε κύριε Ντελάγκε. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Στη συνέχεια